Λοιπόν, έκθεση ΠΑΚ, παράγραφος 1, συμβιβαστική 6, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, δεκτή. Περνάμε τώρα στην 7, καταπίπτουν όλες οι ενδιάμεσες τροπολογίες, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 69. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 69. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 69. Ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Ξαναρχίζουμε λοιπόν. Για την 69. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 34 και μία κατά 50 υπέρ δεκτή. Για την 70 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτό το δεύτερο τμήμα. 71. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έχει αποσυρθεί το 72-73. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. Έχει αποσυρθεί το 76 και το 77. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 78. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 79 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 80 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Φτάνουμε τώρα. Σε δύο τμήματα θα ψηφίσουμε την 81. Το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Το δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 85 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 86. Ποιοι είναι υπέρ. Ζητώ συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος, επανέρχομαι. Έκανα λάθος. Έχοντας απορρίψει το δεύτερο τμήμα του 81, στην ουσία καταπίπτει η 86 και περνάμε στην ψηφοφορία της 88. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 89. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 90. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 91. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έχουμε τώρα τη συμβιβαστική 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 102. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στο 107. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 108. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 110 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τώρα προφορική τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 115. Όχι, γιατί έχει γίνει δεκτή η 3. 117. Είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 118. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έχουμε τη συμβιβαστική στο 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτό. Περνάμε τώρα στη συμβαστική 13. Λοιπόν, 13 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Πηγαίνουμε στην 122. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 126. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 127 υπέρ κατά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 127 ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 54 κατά, 128 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 129 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 15 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 140 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 160 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 169 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 173 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 177 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 178 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 181 υπέρ κατά απορρίπτεται 183 υπέρ κατά δεκτή 182 υπέρ κατά δεκτή 184 υπέρ κατά δεκτή 185 όχι για μια στιγμή όχι αυτή δεν την ψηφίσουμε γιατί έχουμε εγκρίνει την 184 186 υπέρ κατά δεκτή. 187 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 188 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ξεχωριστή ψηφοφορία τώρα για την 190 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της 190. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονική για το πρώτο τμήμα της 190. Ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, και 29 συν 2 κατά απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα λοιπόν της 190 ψηφίζουμε. 191 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά δεκτή. Περνάμε στην 18 υπέρ κατά δεκτή. 19 υπέρ κατά δεκτή. 20 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Δεχτεί. 25 υπέρ, κατά, δεκτή. Συγγνώμη, για το Β στην τροπολογία 12, μόνο το δεύτερο τμήμα εφόσον γίνεται δεκτή συμβιβαστική 2. Το πρώτο τμήμα πρέπει να ψηφιστεί. Θα γυρίσουμε στη 12 λοιπόν. Να ψηφίσουμε και το πρώτο τμήμα της 12. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα της 12. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25. Τροπολογία 25. Α, όχι, ψηφίστηκε 25, συγγνώμη. 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Δεκτό. 28. Υπέρ. Κατά. Δεκτό. 29. Υπέρ. Κατά. Δεκτό. Περνάμε τώρα στην 30. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα της 30. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεν είδα καλά. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της ε, ηλεκτρονικά. Της 30 το πρώτο τμήμα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζετε. Τέλος της ψηφοφορίας. 21 και ε, μία ψήφος 23 υπέρ, 23 και 2 κατά απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα της 30 πάλι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτό. 31 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά Δεκτό. 34 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 35. 35. Ποιοι είναι υπέρ της 35. Α, έχει αποσυρθεί. Δεν το είδα. Συγγνώμη. Προφορική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 36. 37 μάλλον. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 42 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 45 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 45. Καλώς. Ξεκινάει η ψηφοφορία λοιπόν για το 45. «27 κατά, 29 και δύο υπέρ. Γίνεται δεκτή λοιπόν η 45. Έρχομαι στην προφορική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών θα ήθελα στην προφορική του πολύ μια αλλαγή, να αλλάξει το κείμενο και εκεί που λέει διότι διάφορα μέλη δεν έχουν κυρώσει το SAA και επομένω ε, επιβραδύνουν την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προ τη χώρα. Επομένω θα πρέπει τα ε, κρατημέρια αυτά αμιλητή να προβούν στη σχετική κύρωση. Έχει το λόγο η, η, κατά, oh. με, κατά τις τροπολογίες αυτές. Νομίζω πως θα πρέπει να κατονομάσουμε αυτούς οι οποίοι δεν το έκαναν για να τους δώσουμε και ένα κίνητρο να κινηθούν λίγο. Δεν ζητώ λοιπόν να εθετήσουμε την ε, τροπολογία ως έχει για να κατονομάσουμε τους ανθρώπους. Να παραμείνει ως έχει η δική μου, η δική μου προφορική τροπολογία. Bene, allora votiamo l'emendamento orale 2. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική 2 στην προηγούμενη διατύπωση της. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. 48 υπέρ. Κατά. Απορρίπτωσα. 49 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 50 υπέρ κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, δεκτή. 54 υπέρ, κατά, δεκτή. Οι 1, 2 και 3 μαζί. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτέ. 4. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5. Έχει αποσυρθεί. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική παρακαλώ. Ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 48 υπέρ. 50 λοιπόν, άλλοι δύο χωρίς κάρτα. Συγχαρητήρια στη εισηγήτρια. Έχουμε τώρα άλλη μία ψηφοφορία για το μέσο για τη δημοκρατία. Τροπολογία 1. 1, 2 και 3 μαζί ψηφίζονται. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έχει αποσυρθεί 4. Ψηφίζουμε την 9. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. Έχει αποσυρθεί η 5. Ψηφίζουμε τη 10. Ποιοι είναι υπέρ κατά, δεκτή. Η 7 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 και 6 αποσυρθεί, έχουν αποσυρθεί. Η 11 υπέρ, κατά, δεκτή. 12 υπέρ, κατά, δεκτή. 13 υπέρ, κατά, δεκτή. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε. Τέλος της ψηφοφορίας. Σαρανταπέντε συν Δεκτό λοιπόν. Τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίζουμε. Έχετε βάλει όλοι τις κάρτες σας. λοιπόν 46 συν 2, 48 υπέρ, μία κατά. Τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Τώρα. Έχουμε τη γνωμοδότηση για το Πακιστάν. Μία τροπολογία μόνο. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Α, θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για τη μία αυτή τροπολογία. Καλώς. ψηφίζετε. Τέλος. 32 υπέρ, 20 κατά. Τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Λοιπόν, κάποιοι έχετε ξεχάσει τις κάρτες σας μέσα στη θήκη, αλλά δεν ψηφίζετε. Τέλος της ψηφοφορίας. 40 υπέρ, 10 κατά. Συγχαρητήρια λοιπόν. Λοιπόν, τώρα διακόπτουμε τεχνικά για 5 λεπτά. ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να πω ότι έχω απογοητευτεί από αυτή την απόφαση. Βεβαίω και δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και θα πρέπει να μιλήσει κάποιο από την Λιμπέ αλλά σήμερα χάσαμε μια ιστορική ευκαιρία να φανούμε θαραλέοι και λυπάμαι πάρα πολύ λοιπόν θέλω το πέρασμα τη ψηφοφορία, γιατί θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάτι σε σχέση με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Δυστυχώ. θα έπρεπε να είμαστε παράδειγμα προ μίμηση και νομίζω ότι κινδυνεύει η κυρία Μάλστον το όνομά τη να συνδεθεί με ένα τέτοιο κείμενο το οποίο κάνει τόσα, τόσο λίγα πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.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 e poi parla e poi Bene, se gentilmente volete prendere posto possiamo trattare Καθίστε λίγο για να ασχοληθούμε με το θέμα που αφορά την ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην Γάζα μετά την επέμβαση του Ισραηλινού ναυτικού για την αναχέτηση του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον θάνατο κάποιων ακτιβιστών. Πριν περάσουμε στην ανταλλαγή απόψεων, θα ήθελα να πω πως ε, μετά από ρητό αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής ε, Ασφάλειας θα γίνει η συζήτηση αυτή σε δύο χωριστά τμήματα. Παρουσία του κυρίου Πρέσβη, του κυρίου Κούριελ και του Φερνάντε Τσάριας. Κατόπιν θα έχουμε μία πρώτη φάση μετά την παρέμβαση του πρέσβη του κυρίου Φερνάντες Άριας ε, που θα αφορά την ε, θέση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης μετά την δήλωση της υπατής εκπροσώπου και μετά θα ακολουθήσει η παρέμβαση του πρέσβη του κυρίου mm. Κούριελ και βεβαίως τα δικά σας σχόλια και αιτήματα. Δεν επειδή δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, θα αφήσω όλο τον χρόνο που απαιτεί Πού απαιτείται. Στους ε, συναδελφούς και στους δύο μιλητές μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να δώσω τον λόγο στον πρεσβευτή, στον κύριο Φερνάντες Άριας. Παρακαλώ κύριε πρεσβευτά. La ε, ringrazio, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. ευχαριστώ που με καλέσατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να σας ε, εξηγήσω περί τίνος πρόκειται, τι έχουμε κάνει ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν των χθεσινών συμβάντων. Όπως αναφέρατε, είχαμε αυτό το πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο έχει αποπειραθεί να προσεγγίσει τη λωρίδα της Γάζης. Επιτρέψατε μου τώρα να σας ε, αναφέρω ότι σήμερα βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας την υψηλή εκπρόσωπο. Για να σας πω επομένως τι επαφές είχαμε χθες και σήμερα. Επίσης, να πούμε δύο λόγια σε σχέση με το τι πρόκειται να ακολουθήσει τα όσα έγιναν. Η Κάθριν Άστον μόλις λίγες ώρες κατόπιν των όσων έγιναν ήρθε σε επαφή με όλους τους εμπλεκομένους με τον υπέξ του Λιβάνου και σήμερα το πρωί τον κύριο Φαγιάτ της ε, Παλαιστινιακής Αρχής. και τον ε, υπέξ του Ισραήλ, τον κύριο Λίμπερμαν. Και χθε ήρθε επίση ε, έγινε συνεργασία με τον επικεφαλή του Διτεργογραφείου. Οπότε, γι' αυτό και προσπάθησε υψηλή εκπρόσωπο να γίνει μια συνεδρίαση, ούτως ώστε να συνταχθεί μια δήλωση για να συγκεράσουμε όλες τις ε, απόψεις και να δημορφωθεί έτσι μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα όσα έγιναν. Πρόκειται για αντίδραση ταχεία και ε, πρόκειται για μια προσπάθεια του να υπάρξει κοινή θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ε, έντονη η αντίδραση, βεβαίως αυτό είναι φυσιολογικό, διότι πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρό και τραγικό συμβάν. Νομίζω ότι έχετε λάβει το κείμενο της ε, δήλωση και ίσω οι περισσότεροι το έχετε διαβάσει. πάντω πάντως κάποια άλλα στοιχεία εδώ. Πρώτα-πρώτα καταδικάζουμε την απώλεια ανθρώπινη ζωή. Και επίσης συλληπούμεθα τι οικογένειε των θυμάτων. Καταδικάζουμε την χρήση βίας που οδήγησε σε τόσα θύματα. Επίσης, ζητούμε να αρχίσει μια έρευνα αμερόληπτη και πλήρης για τις συνθήκες του επεισοδίου. Τώρα υπάρχουν τα εξής άλλα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να προσθέσουμε. Πρώτα-πρώτα ζητούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην έχουμε κλιμάκωση της βίας και των σχετικών επεισοδίων. Επίσης, ζητούμε από τις Ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν πλήρη εξυπηρέτηση των όσων έχουν εμπλακεί σε αυτό το επεισόδιο, πλήρη πρόσβαση στις προξενικές τους αρχές. Και σε σχέση με τον αποσμό της Γάζας επίσης ζητούμε αυτό να αρθεί για άλλη μια φορά. Αυτή ήταν μια αντίδραση επομένω, η οποία έγινε στη συνέχεια της πρώην δήλωσης και ακολουθήθηκε από την δήλωση Λαυρόφ στο Ροστόφ γιατί εκεί είχε γίνει η συνάντηση κορυφής ΕΕ Ρωσίας. Έχουμε επίσης και τη δήλωση του πρόεδρου την σήμερα το πρωί. Σειρά άλλων δηλώσεων επίσης έχουν γίνει χθες ε, στον ΟΗΕ. Μετά από αυτή την πρώτη αντίδραση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διπλωματικές και πολιτικές συνέπειες. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. θα υπάρξει πίσω προς πανσενίους, να αρχίσουν έμεσες επαφές, πολύπλοκες δημοτικές προσπάθειες και φοβούμε ότι επίσης θα ενταθούν ε, ήδη ε, δύσκολες εκεί σχέσεις. Επίσης ε, ήδη έχουμε την αντιπαλότητα με την Τουρκία και εκεί θα έχουμε επιδείνωση των σχέσεων. Ήδη υπάρχει επομένω στροφή προς τα χειρότερα και θα πρέπει και αυτό να εξομαλυνθεί το συντομότερο. Επίσης, έχει υπάρξει πίεση και προς την Αίγυπτο να ανοίξει τα περάσματα προς τη Γάζα. Και επομένως θα πρέπει εμείς να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις συνέπειες. Είδαμε την κλιμάκωση, ε, θα μέσα μας και ενημέρωση και ε, συλλαλητήρια, δηλώσεις και γι' αυτό και εμείς είπαμε προς ε, όλους να αποφύγουν την κλιμάκωση και τη χειρότερη ένταση. Όλοι μας θα κάνουν, πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούμε σε αυτή την κατεύθυνση για να συνεχιστούν οι επαφές ε, προσέγγισης. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μην ξεχνούμε επίσης ότι ο τελικός στόχος εδώ είναι να πρετανεύσει η ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εκπροσώπων της έχει συνεχώς επαφή με το κουαρτέτο. Ψήρα επαφών χθε και σήμερα. Συμφώνησε το κουαρτέτο ε, είπαμε ότι είναι και επαφή στο Ροστόφ μεταξύ Λαυρόφ και Άστον Και είπαμε το σωμότερο δυνατόν ίσω και τον Ιούλιο να υπάρξει και άλλη επαφή μεταξύ ε, των τον Λαυρόφ και Άστον τον Ιούλιο για να ληφθούν υπόψη και να συνεχιστούν τα όσα ελέγχθησαν χθες και περιέχονται σχετική δήλωση. Να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι μακρόπνες, πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες. Υπάρχουν και κάποια συμπεράσματα που μπορούμε να αντιλήσουμε από τα όσα έγιναν. Πρώτα-πρώτα, κάτι το οποίο ξεκάθαρα περιέχεται στη χθεσινή δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχθεί ε, τη συνέχιση του αποκλεισμού τη Λωρίδα τη Γάζα. Είναι κάτι το απαράδεκτο, είναι κάτι το αντιπαραγωγικό. Θα πρέπει επίσης να ανοίξουν το σχετικά περάσματα πρόσβασης υπό εποπτεία παρακολούθηση. Όπως ξέρετε εμείς έχουμε μακρά δέσμευσε, ούτως ώστε να ανοίξει η περιοχή, το πέρασμα της Ράφα. Υπάρχει αποστολή, έστω και σε αδράνεια εκεί και επομένως μόλις θα βάλει μπλεκόμενοι θα ανοίξει το πέρασμα. Θα πρέπει να βρεθεί μια λειτουργική λύση για το πρόβλημα της Γάζας και πρέπει να υπάρξει επομένω μια βαθιά αλλαγή στην πολιτική προ τη Γάζα. Είναι πολιτικό το πρόβλημα και άρα επιδέχεται λύση πολιτική. Κατόπιν αυτών των επεισοδίων δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να γνωρούμε τη Γάζα. Εδώ τελείω κύριε Πρόεδρε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πέζη. Ο κύριος Αλαφράγκα δύο λεπτά παρακαλώ. Πρώτα πρώτα ε, ευχαριστώ τον ε, ε, εκπρόσωπο της κυρίας Άστον που τόσο γρήγορα ήρθε εδώ και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό θα πρέπει να σας εκφράσω το ότι επίσης και εμείς καταδικάζουμε την απώλεια ανθρώπινης ζωής και πέραν των όσων μας, μας είπαν παρά το τις εξηγήσεις του, του, του πρεσβευτή δεν είναι δυνατόν να καταδικάσουμε ε, αυτές τις ενέργειες που προέρχονται από ένα από τους πιο σύγχρονους στρατούς του κόσμου. Έχασαν λοιπόν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι και όταν έχουμε τέτοια γεγονότα θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε ποιες είναι οι αιτίες και ποια είναι τα αποτελέσματα. Η ε, αιτία είναι αυτό το εμπάργκο, αυτός ο αποκλεισμό εις βάρος του, των κατοίκων της Γάζας, άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Για κάποιες, ε, για, κάποιες ενέργειες μπορεί να έχουν τέτοιου είδους ε, συνέπειες. Να, μας τα είπε τώρα ο εκπρόσωπος της ε, κυρίας Άστον. Έχουμε επομένως τώρα επιδείνωση της προσπάθειας για την ειρήνη, έχουμε απομόνωση του Ισραήλ, έχουμε την, ε, την αλλαγή της, της, της πολιτικής των ΙΠΑ, την, την επιδείνωση των σχέσεων και απόσυρση του πρεσβευτή της Τουρκίας και όλοι επομένως μπορούμε να διαπιστώσουμε και τις τόσο σημαντικές ε, συνέπειες που δεν μπορούν παρά να επηρεάσουν τη διεθνή σκηνή. Για πέστε μας παρακαλώ, πόσοι Ευρωπαίοι τώρα βρίσκονται εκεί, πόσοι έχουν εμπλακεί. Είπατε ότι ζητήθηκε προσβασιμότητα στα προξενία και στις προξενικές υπηρεσίες, αλλά τι, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική μας. Μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε τον χαρακτηρισμό της Χαμάς που βρίσκεται στη μαύρη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων για εμάς τους Ευρωπαίους. Κύριε Σαλαβράκη, ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η επόμενη παρέμβαση Μούνιτς. Δύο λεπτά. Ευχαριστούμε την Προεδρία, ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της της εξωτερικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε αυτό το οποίο έγινε είναι παράγον αστάθειας για την περιοχή. Καταλήτης αστάθειας γιατί πάρα πολλοί θεωρούμε ότι αυτό το οποίο έγινε είναι δυσανάλογη χρήση βίας για την προστασία αυτού του αποκλεισμού και βαριά παράβαση του διεθνούς δικαίου και ταυτόχρονα πράξη επίθεσης. Και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης ε, υπέστησαν παραβιάσεις. Το Ισραήλ επομένω γίνεται κράτος το οποίο για να προστατεύσει την ασφάλεια προβαίνει σε πράξεις πειρατείας. Θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για όλα αυτά. Θα πρέπει επίσης να δοθεί νέα όθηση στην ειρηνευτική διαδικασία. Να μπορέσουμε αυτή την προσπάθεια να την πλαισιώσουμε με, με, ό,τι γίνεται το νωρίτερο δυνατόν. Και θα πρέπει να ζητηθεί το τέλος του εμπάργου που δεν είναι εμπάργου, που είναι αποκλεισμό της Λόριδας της Γάζας. Αυτό είναι κάτι που πάρα πολύ απαραίτητο να γίνει. Κυρία δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές ε, την αποδοκιμασία της ε, για τον αποκλεισμό της Γάζας για ανθρω... και έχει ζητήσει να έρθει για ανθρωπιστικούς και για πολιτικούς λόγους και τα τραγικά γεγονότα των προηγούμενων ημερών έδειξαν ακόμη μία φορά πως η κατάσταση πράγματι δεν μπορεί να συνεχιστεί ως ε, έχει. Γιατί έχει, βλέπετε, τέτοια αρνητικά αποτελέσματα. Αυτονόητο είναι πως η δική μου ομάδα καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ στον ε, Λίσκο. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω εάν μπορεί να εξακριβωθεί το εάν ε, όντως η επίθεση έγινε στα διεθνή ύδατα. Ε, κάτι το οποίο βεβαίως σύμφωνα με τη διεθνές θα την καταστήσει ακόμη χειρότερη. Κιλ Νίλσεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Μόλις επιστρέψαμε από τη Λωρίδα της Γάζα, ήμουν με τους συναδέλφους εκεί. Το 2009 μου είχε στερήσει το Ισραήλ τη δυνατότητα να πάω. Εν πάση περιπτώσει αυτή τη φορά πήγαμε μέσω της Αιγύπτου. Πρώτη φορά πήγα στην Αίγυπτο. Και κατάλαβα γιατί το Ισραήλ δεν ήθελε να πάμε στη Γάζα. Ήταν απλό. Μιλάμε για ένα γκέτο. Η ζωή σε αυτό το γκέτο είναι ανυπόφορη. Είναι σκάνδαλο το να διατηρούνται σε τέτοια κατάσταση όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάτω, ε, το 50% είναι κάτω των 20 ετών και δεν μπορεί καν να τους κατηγορήσει κανείς ότι ψήφισαν λάθος γιατί δεν ψήφισαν. Το μοναδικό δικαίωμα που έχουν όλοι αυτοί στη Γάζα είναι το να επιβιώνουν, δεν έχουν το δικαίωμα στη ζωή. Η τραγωδία την οποία βιώσαμε με, αυτή, με αυτό το στολίσκο για την ειρήνη ε, είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι. Νιώθω κι εγώ γιατί είμαι υπεύθυνοι. Οι κυβερνήσεις, η πολιτική, η ένωση. Δείχνουμε ένα τεράστιο, ε, μια τεράστια έλλειψη πολιτικού θάρρους απέναντι στο πρόβλημα της Παλαιστίνης και της Γάζα. Δεν λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις, δεν λαμβάνονται γενναίες αποφάσεις. Γι' αυτό οι πολίτες παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Αυτό είναι σκανδαλώδες αυτή η διαδικασία του μποϊκοτάζ που αναπτύσσεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Γιατί αυτό, γιατί δεν είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε το ότι στα προϊόντα τα οποία εισάγουμε να μην υπάρχουν προϊόντα από κατεχόμενα εδάφη, γιατί δεν διασφαλίζουμε την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων μας. Επιδεικνύουμε μια τεράστια έλλειψη πολιτικού θάρρους. Και γι' αυτό οι πολίτες παίρνουν πρωτοβουλίες. Ο θάνατος αυτών των ειρηνιστών, ο θάνατος αυτών των ανθρώπων, ελπίζω αυτή τη φορά να μας οδηγήσει στο να πούμε ότι ας αλλάξουμε πια άποψη και ας θέσουμε τέλος την ατιμορρησία του κράτους του Ισραήλ. Τάνοκ δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Οπωσδήποτε η ομάδα μας λυπάται για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών, αλλά είναι ξεκάθαρο πως ο Ισραηλινός στρατός δεν σκόπευε εξ αρχής να χρησιμοποιήσει θανάσιμη βία και στα πέντε από τα έξι πλοία κατάφεραν ειρηνικά να τα εκτρέψουν και να πάνε σε ένα λιμάνι στην επικράτεια τους. Επίσης είχε προειδοποίησει την IHH μια Ισλαμική ανθρωπιστική οργάνωση που οργάνωσε την όλη εκδήλωση πως δεν θα δεχόταν το σπάσιμο του αποκλεισμού όσο η Χαμάς εξακολουθεί να εκτοξεύει βλήματα κατά πολιτών και να δέχεται βλήματα. Το Ισραήλ θεωρεί πως ο αποκλεισμός είναι νόμος, εγώ τώρα δεν ξέρω το δίκαιο της θαλάσσης, αλλά δεν ε, εμποδίζει ανθρωπιστική βοήθεια διαξηράς. Μέχρι και η Αίγυπτος έχει κλείσει τα σύνορά της στην ξηρά ακριβώς από όταν ανέλαβε την κυβέρνηση Χαμάς και χρησιμοποίησαν οι στρατιώτες του Ισραήλ ε, θανατηφόρο βία μόνο όταν απειλήθηκε η ίδια τους η ζωή από ράβδους, μαχαίρια και άλλα τέτοια. Είναι δικαίωμά τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αλλά αν χρησιμοποίησαν δυσανάλογη βία, ζητώ να ερευνηθεί αυτό πλήρως από τον στρατό του Ισραήλ και βεβαίω να υποστούν τα όσα προβλέπει ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας. Αλλά είναι σαφές πως η αποστολή είχε στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό ως χειρονομία, όχι να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια. Και έχουμε ξεκάθαρα τώρα μαγνητοσκοπημένες εικόνες ανθρώπων που φωνάζουν τζιχάτ και εντιφάντα και υποδείχνουν ότι είναι ειρηνιστές. Η παρουσία δε γυναικόπαιδων στα πλοία αυτά γνωρίζοντας πώς θα μπορούσε να ξεσπάσει η βία είναι επίσης απράδεκτη και την καταδικάζουμε. Εμείς στο κόμμα μας λυπούμεθα για την απώλεια εννέα αθώων ζώων και οποιοδήποτε έδρασε εκτός νόμου πρέπει να λογοδοτήσει αλλά όπως σας είπα το Ισραήλ αντιμετωπίζει κίνδυνο για την ύπαρξή του και δεν μπορεί να ρισκάρει την διέλευση όπλων προς την Γάζα, προς την Χαμάς που θα σας επενθυμίσω είναι μια τρομοκρατική οργάνωση σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ισραήλ και η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή αντιμετωπίζουν απειλή από την Χαμάς. Ευχαριστούμε. Μέιερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς πρώτα απ' τα δημόσια θα πρέπει εδώ να τιμήσουμε όλους όσους αθώοι, ακτιβιστές έδωσαν τη ζωή τους που ήθελαν να πάνε και να φέρουν αυτούς τους χίλιους τόνους της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λόριδα της Γάζας. Θα πρέπει επομένως να κάνουμε έναν απολογισμό του τι έγινε και έναν καταλογισμό των ευθυνών για αυτό το έγκλημα του της κυβέρνηση του Ισραήλ που έχει βάψει τα χέρια της με αίμα αθώων. Δεν είναι δυνατόν αυτό να μείνει ατιμόρυτο. Η ΔΕ Ένωση έχει, έχει και με το παραπάνω τρόπο ούτως ώστε να βοηθήσει και η πολιτική αλλά και η ποινική ευθύνη να αποδοθεί προς την κυβέρνηση του Ισραήλ γιατί πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου από αυτές που έχει συνηθίσει η Ισραηλινή κυβέρνηση η οποία προσυπέγραψε την συνθήκη της Νάπολης αλλά δεν τηρεί τα υπεσχημένα και έτσι δεν κάνει τίποτα ώστε να μπορεί να έχει γείτονα ένα Παλαιστινιακό κράτος. είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση, θα πρέπει επομένω να γίνει ψήφισμα και συζήτηση στο Στρασβούργο να γίνει αυτό και να ολοκληρωθεί ένα ψήφισμα και όλες οι πολιτικές ομάδες να τοποθετηθούν λέγοντας τι είδους καταδίκη θα πρέπει να γίνει και να μην μείνει το έγκλημα ατιμόρυτο. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, εάν δεν είναι δυνατόν να, να κάνουμε τίποτε άλλο θα πρέπει να ζητήσουμε την, την, την τήρηση των υπεσχημένων. Έχουμε συμφωνία με το Ισραήλ, υπάρχει μια σχετική ρήτρα και άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να παγώσουμε την συμφωνία σύνδεσης. Γιατί δεν το ζητούμε αυτό, γιατί δεν έχουμε πιο δυναμική τοποθέτηση όσον αφορά την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε 400 πολιτικούς κρατούμενους ε, τώρα. Έχουμε 10... 10 περίπου και πολύ παραπάνω νεκρούς. Ε, δεν δε, δε δικαιολογούν αυτά τα νούμερα μια άλλη αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς αυτό θα, θα κάνουμε προς τα εκεί, γιατί θα κινηθούμε με το κείμενο το οποίο πρόκειται σαν δήλωση να συντάξουμε. Ωραία, πρώτος γύρος των παρεμβάσεων, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Φερνάντες έχει τώρα το λόγο για να απαντήσει σε αυτά τα που ελέγχθηκαν στον πρώτο γύρο. Και όταν είναι ο κύριος Πρέσβης. Ευχαριστώ. Ναι, έχουμε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν θέλω να πω τίποτα για τα σχόλια, απλώς για τις ε, ερωτήσεις που όπως σωστά είπατε ε, μερικά θέματα είναι θέματα του κύριου Πρέσβος. Ο κύριος Αλαφράγκα ερωτά πόσοι είναι οι Ευρωπαίοι που τώρα όπως γνωρίζουμε κρατούνται βρίσκονται τέλος στο Ισραήλ. Δεν έχουμε πλήρης ακριβής πληροφορίες Υπήρχαν ε, κάποιοι Ευρωπαίοι που είχαν επιβεί αυτών των, πλοίων οι οποίοι τελικά από το Ασδότ το λιμάνι ε, πήγαν στην Μπερσεβά κάποιοι από αυτούς επαναπατρίστηκαν ευθύ αμέσω. άλλοι όμως προτιμήσανε να μην δώσουν τα στοιχεία τους να μην κάνουν τις σχετικές δηλώσεις θεώρησαν ότι αυτό είναι κομμάτι κάποιας παθητικής αντίστασης. Αυτά τα στοιχεία έχουμε κατόπιν των επαφών που είχαμε με το Τελαβίβ και συνεργαζόμαστε με τις εκεί δικαστικές αρχές σε σχέση με την Ισραηλινή νομοθεσία που ρυθμίζει την νόμιμη και παράνομη μετανάστευση στη χώρα. Έχουμε τώρα τις τελευταίες ώρες κάποιες φρέσκες πληροφορίες. Τις τελευταίες τέσσερις ώρες μας έχουν πει για περίπου 50 Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι κρατούνται στο Ισραήλ, οι περισσότεροι στη Βερσεβά και περίπου άλλοι 10 έχουν ή πρόκειται άμεσα να επαναπατριστούν και έχω και στα αριθμικά στοιχεία αναεθνικότητα να σας ενδιαφέρει. Όμως υπάρχουν και κάποιες χώρε που δεν έχουν και διπλωματική αντιπροσωπεία ή τέλο πάντων δεν μπορέσανε να βρουν τα σχετικά στοιχεία. Οπότε έχουν απλώ κάποιε πιθανολογήσει. Είναι σημαντικό επομένω αυτό το οποίο ζητήσαμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση από τι Ελληνέ Αρχέ, ώστε να, επιτρέψουν την πρόσβαση των, των Ευρωπαίων στι προξενικέ του ε, αρχέ. Τώρα για τη Χαμά, κύριε Σαραφράγκα, συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρεί τη δέσμευσή τη ε, σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και επίσης ε, του κορτέτους 19 Μαρτίου όσον αφορά το ότι θα πρέπει να πληρεί η Χαμάς πρώτα από την αναγνώριση του Ισραήλ σαν προϋποθέσεις να καταδικάσει τη βία και επίσης να σεβαστεί τις ε, συμφωνίες που, ε, με τις οποίες έχει συνάψει. Αυτές ήταν προϋποθέσεις και αρχές της Ένωσης που δεν έχουν αλλάξει. Τώρα, η κυρία Νέιτς. Ερώτα. Αν η επίθεση έγινε σε Μα αυτό αναφέρουμε και στη δήλωσή μας ότι πρόκειται για διεθνή τα σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε. Όπου ε, τα σκάφη ή τέλος πάντων το βασικό το τουρκικό σκάφος βρισκόταν περίπου 62 ναυτικά μίλια μακριά από την ζώνη που έχει αποκλειστεί. 80 περίπου 70 με 80 ναυτικά μίλια από τις Ισραηλινές ακτές της Λωρίδας της Γάζας, του Ισραήλ, ανάλογα με ποιες παραμέτρους επικαλείται κανείς. Γι' αυτό και μιλούμε για διεθνή είδατα. Γιατί η Γάζα σας τα είπα, δεν έχει αλλάξει τίποτα στην πολιτική μας και αν υπάρχει κάτι καλό που βγαίνει από αυτά τα τραγικά γεγονότα είναι το ότι η κατάσταση στη Γάζα τώρα είναι πάλι κάτι που έχει διεθνοποιηθεί. Δεν μπορώ να πω αξιολικές κρίσεις, αν είναι για καλό ή για κακό, αλλά πάντως μη συνεχίζουμε πιστεύω ότι θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να ασχοληθεί με τη Γάζα. Και αυτό και θα γίνει με μεγαλύτερη σοβαρότητα από το και στο εξή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες, κύριε Πρέσβη. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Πρέσβη, τον κύριο Κούριελ. Thank uh, κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, συνάδελφοι της Προεδρίας και του Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους σας και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Τα πρόσφατα γεγονότα δεν ήταν εύκολα για κανέναν να πω πως πρώτα απ' όλα εμείς στο Ισραήλ λυπούμεθα για την απώλεια ζώων. Φαντάζομαι πως παρακολουθήσατε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Στο χρόνο που μου δώσατε μάλλον δεν θα μπορέσω να καλύψω όλα τα στοιχεία, θα προσπαθήσω να αναφέρω κάποια από αυτά που είναι η βάση της θέσης και των διλημάτων του Ισραήλ. Να ξεκινήσω λέγοντας κάποια από τα λόγια που είπε χτες το βράδυ ο πρόεδρος ο κ. Σίμων Πέρες. Η Χαμάς, είπε, αποφάσισε να εμποδίσει την ειρήνη μεταξύ των Παλαιστινίων και το Ισραήλ. Το Ισραήλ εκένωσε τη Γάζα η Χαμάς τη μετέτρεψε σε μια βάση επίθεσης κατά του Ισραήλ και εκτόξευσε πάνω από 10.000 βλήματα κατά Ισραηλινών πολιτών. Συνεχώς αποκτά και με λαθρεμπόριο όπλα και βλήματα στη λορίζα της Γάζας μέσω τούνελ και διαθάλασσης Η Χαμάς γνωρίζει πως μπορεί να ακολουθήσει την ίδια πορεία με την Παλαιστινιακή Αρχή και να φέρει ευημερία και ειρήνη στο λαό της. Όμως επιλέγει την τρομοκρατία αντευτού. Ο συνάδελφος ο Ισπανός πρέσβης ανέφερε τα βασικά στοιχεία του κουαρτέτου που είναι το κεκτημένο των συνομιλιών τα οποία η Χαμάς το αρνείται. Δεν τους ζητάμε να αναγνωρίσουν το Ισραήλ, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει. Ζητάμε, αλλιώ δεν υπάρχει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το Ισραήλ δημοκρατικό κράτος, εδώ πέρα συνεχίζω να διαβάζω τα λόγια του Πρόεδρου Πέρες, το οποίο έχει στόχο να ε, προστατεύει τις πολίτες του, δεν μπορεί να δεχτεί την αύξηση πλοίων που δεν έχουν ελεγχθεί στην Γάζα. Η βίαιη και ο βίος και προκλητικός στολίσκος ε, είχε στόχο την στήριξη της Χαμάς, κατά το οποίο σημαίνει τη στήριξη της τρομοκρατίας και την άρνηση της ειρήνης. Εδώ πέρα τελειώνουν δηλώσεις του Πρόεδρου. Το άλλο ζήτημα που ήθελα να δείξω είναι το ζήτημα του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, μιας οργάνωσης, όπως αναφέρθηκε, που είναι στον κατάλογο της τρομοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον συνεχώς μπαίνουν όπλα στη Γάζα και διαδαλάσεις, ο ναυτικός αποκλεισμός είναι θεμητό και αναγνωρισμένο από το Διεθνές Δικαιομέτρο και μπορεί να εφαρμοστεί στην θάλασσα και στα διεθνή ύδατα. Συνεπώς το Ισραήλ ήταν εντός του διεθνούς δικαίου όταν προσπάθησε να εμποδίσει την πορεία του στο Με την αδειά σα θα ήθελα να δώσω στον πρόεδρο της Επιτροπής μια σύντομη νομική ανάλυση που υποστηρίζει αυτά που λέω για να σας την μοιράσει γιατί είναι εύκολο να λέμε τις λέξεις διεθνές δίκαιο αλλά εδώ, σε αυτή την περίπτωση, το Ισραήλ βρίσκεται εντός των δικαιωμάτων του. Όλοι γνωρίζετε από τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες σε διάφορους διάβλους και σε όλα τα επίπεδα και με δημόσιες δηλώσεις ξεκαθάρισε το Ισραήλ θέση του έναντι αυτού του στολίσκου και προσέφερε στους διοργανωτές την μεταφορά του ανθρωπιστικού φορτίου μέσω του λιμανιού του Ασντόντ αφού περάσει, αφού εξεταστεί. Οι άνθρωποι στα πλοία αυτά ισχυρίστηκαν πως έχουν 10.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλω να γνωρίζετε, έτσι για να έχετε υπόψη την αναλογία, πως κάθε εβδομάδα περνάνε 15.000 τόνοι ε, μέσω του Ισραήλ για την Γάζα. Μπορώ να σας πω με λεπτομέρειες ε, το τι μπαίνει στη Γάζα και με ποιο τρόπο. Παρά τις προσπάθειες του Ισραήλ, οι οργανωτές από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρονταν να οργανώσουν μια βίαιη και προσχεδιασμένη πρόκληση. Οι οργανωτές ξεκαθάρισαν πως βασικός τους στόχος ήταν ο ναυτικός αποκλεισμός. Η Γκρέτα Μπερλίν, εκπρόσωπος του Στολίσκου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως η αποστολή αυτή δεν αφορά ανθρωπιστικά εφόδια, είναι για να σπάσει η Ισραηλινή πολιορκία επιβιβαζόμενοι σε ένα από τα έξι πλοία, οι Ισραηλινοί στρατιώτες υπέστησαν επίθεση από όχλο υπέρτερο σε αριθμό που χρησιμοποιούσε ρόπαλα. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες ήταν οπλισμένοι με όπλα για την αυτοάμυνά τους. Με χρώματα που τους επιτέθησαν λοιπόν με ρόπαλα, σφεντώνες και άλλα όπλα και απειλούνταν η ζωή του. Δύο Ισραηλοί στρατιώτε τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τρει άλλοι είναι σε... τραυματίστηκαν λεφρά. Όλα τα θύματα είναι στο Ασντόντ. Στα υπόλοιπα πλοία επιβιβάστηκαν χωρί πρόβλημα. Ζήτησα από τη γραμματεία να μου επιτρέψει να σας δείξω μια φωτογραφία της απόπειρας αυτής λιντσαρίσματος κατά τη διάρκεια επιβίβαση στο πλοίο.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 Οχι, με Είναι απόλυτα. Είπε. Είτα λοχαδεύαλα κας. Μετά. Παρακαλώ. Μετά, μετά τον κύριο Πρέσβη. Να, να τελειώσει και θα έχετε όλη χρόνο να μιλήσετε. Παρακαλώ, τελειώστε κύριε Πρέσβη. You can see in the photo the... Είδατε τα όπλα τα όπλα που πιάσαμε χτες. Όχι. Ε, πώς, πώς επαληθεύονται αυτές οι εικόνες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσαν να πούνε ψέματα. Λοιπόν, θα έχετε το λόγο όταν σας τον δίνω εγώ. Λοιπόν, θα κλείσει ο κύριος Πρέσβης και μετά εσείς θα έχετε το χρόνο να αμφισβητήσετε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Θα τελειώσω σύντομα. Κυρίες και κύριοι, τι ειρηνιστές έρχονται οπλισμένοι με ρόπαλα και μαχαίρια. Μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρω πως δεν είναι μία ομάδα μόνο. Είναι άνθρωποι από πολλές χώρες και είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίζουμε ως ένα, αλλά η πλειοψηφία, η ηγεσία αποκαλούν αυτούς υπεραστητέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν μιλάνε όταν εσκεμμένα στοχεύει Ισραηλινού πολίτε η Χαμά και για τι ακρότητε ε, του καθεστώτο Χαμά στην ίδια τη Γάζα που έχει συντρίψει την αντιπολίτευση, τα ανεξάρτητα ΜΜΕ και έχει φυλακίσει εκατοντάδε αντιφρονούντε. Δεν ξέρω αν τα είδατε αυτά όταν ήσασταν στη Γάζα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πρόκειτο για ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή. Ήταν μια πρόκληση που τελείωσε τραγικά. Τα γεγονότα εκτιλήσονται και θα συνεργαστεί το Ισραήλ πλήρως με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις προξενικές πτυχές για τους διάφορους επιβάτες των πλοίων. Η ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρεται στη Γάζα μετά τους απαιτούμενους ελέγχους να τελειώσω λέγοντας πως πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε στο πώς θα προωθηθεί η ειρήνη μεταξύ ημών και των Παλαιστινίων και πολλοί στηρίζουν τις ε, συνομιλίες από τους συνεγγείς που ξεκινήσαν πρόσφατα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αν θεωρεί ο κύριος Πρέσβης πως αυτές οι εικόνες θα με πείσουν, ε, έχει τελείως λάθος. Αυτό το οποίο είδα εγώ δεν είναι όπλα. Είναι μαχαίρια που μπορούν να φτιάξουν και σάντουιτς. Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Και όπλα να ήταν. Και όπλα να ήταν. Δεν θα έπρεπε να σκοτώσετε ανθρώπους σε αυτό το πλοίο. Κύριε Πρόεδρε, στη Γάζα ζουν άνθρωποι, οι φτωχότεροι νέοι άνθρωποι, σε άθλιες συνθήκες και με την πολιτική σας τους οδηγείτε στα χέρια της Χαμάς. Και αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάνει ωραίες δηλώσεις και λέτε πως πρέπει να τελειώσει ο αποκλεισμό. Αν δεν σταματήσει τι θα κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο ε, ερώτημα. Προς την Κομισιόν. Δεύτερον, η έρευνα που πρέπει να γίνει. Θα το κάνετε αυτό, κύριε Πρέσβη, θα συνεργαστείτε με την έρευνα. Ή θα γίνει ό,τι και με την έκθεση Goldstone. Και τα ζητήματα της ε, προξενικής πρόσβασης έχουν ρυθμιστεί. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω. Παντσέρι για δύο λεπτά. Εγώ πρόεδρε. Θεωρώ δεν μπορούμε να απομονώσουμε αυτό το θέμα σαν να ήταν ένα μόνο επεισόδιο γιατί εδώ πέρα υπάρχει σύνδεση με το απότερο παρελθόν. Ούτε θα πρέπει να περιοριστούμε στο θέμα των αναγενώσεων. Έχουμε το θέμα της αποστολή εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εδώ. Το πώς δηλαδή θα έρθουν οι φραγμοί προς την ειρήνευση και νομίζω ότι έτσι όπως έγινε η ιστορία της Γάζας έχουν ευθύνε και η ΜΕΝ και η ΔΕ ε, δεν λήφθησαν οι απαραίτητε ε, ενέργειε τόσο να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια. Άρα θα πρέπει να πούμε στου Ελληνού ότι είμαστε ε, έτοιμοι να, να βοηθήσουμε όπου χρειάζεται και δεν κατέστη δυνατό να μπορέσει να πάει τελικά αντιπροσωπεύει του Κοινοβουλίου στη Γάζα. Αυτό είναι ηλίθιο από πλευρά πολιτική, ε, επιτρέψτε να σα πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι η γραμμή πορεία θα πρέπει να την συνεχίσουμε. Έτσι θέτουμε εν κινδύνο την όλη ειρηνευτική διαδικασία. Γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε με τα πλοία και το τι υπέστησαν αυτοί οι άμαχοι αυτοί οι πολίτες. αφελώς επέβησαν πάντως για ε, αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά τα πλοία. Θα πρέπει να γίνει φυσικά μια ανεξάρτητη έρευνα, να δούμε πώς χάθηκαν αυτές οι ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο σπλούνται και την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αποδείξετε ότι δεν είμαστε αδιάφοροι, αλλά το ότι μπορούμε να αντιδράσουμε δυναμικά και ότι θα πρέπει να αρχίσουν οι επαφές άμεσα για να υπάρξει κάποια συνέχεια και θα πρέπει να σταματήσουμε να αναβάλουμε την ανάληψη ενεργειών θα πρέπει να προβάλλουμε επίσης ότι, ότι, ότι πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να κάνουμε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει το σύντομο. Κύριε Παντζέρη, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Βάγγελ, έχετε τώρα για δύο λεπτά. Ισραήλ ραωνά τα κόκο τραωνά, το κεριμά Ευχαριστώ. Το Ισραήλ ε, δρά έτσι γιατί έχει την αίσθηση πως δεν έχει κανένα φίλο στον κόσμο και είναι απομονωμένο και μόνο το κακό του θέλουν όλοι. Δυστυχώς πριν ε, πάει η αντιπροσωπεία στην Παλαιστίνη. Υπήρξαν απόπειρε εδώ μέσα εντός ε, του Κοινοβουλίου να παρουσιαστούν τα μέλη της αποστολής ως άτομα τα οποία αδικούν το Ισραήλ. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ κακό και αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση. Τίθε όμως το ερώτημα πώς απαντάμε στο αίσθημα αυτό απομόνωσης του Ισραήλ. Είναι υποχρέωση του δημοκρατικού κόσμου να δώσει στο Ισραήλ την αίσθηση της ασφάλειας. Και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα από τους γείτονες του Ισραήλ. Και αυτό θα γίνει μέσω... Και αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από τα δύο κράτη, το Ισραηλινό και το Παλαιστινιακό, που θα συνεπάρχουν ειρηνικά. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην Γάζα. Το είδαμε αυτό και θα το συζητήσουμε. Υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άποψή μου, το οποίο είναι η κατάσταση στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Το ότι δηλαδή συνεχίζονται οι Ισραηλοί επικισμοί, το γεγονός πως ε, έχουμε ένα κοινικό apartheid κάτι το οποίο θα δημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα που, το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στη Γάζα. Ευχαριστώ, Ζωλή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας πω την Παρασκευή τι είδαμε στη Γάζα. Ήμασταν εκεί και συναντήσαμε τον υπεύθυνο γιατί είχε δει τη βία, τη βία που ασκεί το Ισραήλ και είχε δει τι βία υφίστανται, τι εκφοβισμό οι κάτοικοι της Γάζας. Δεν μπορούν να ψαρέψουν σε αυτά τα τρία μίλια που θα μπορούσαν γιατί τους έχει συρρυκνώσει την σχετική ζώνη ελεία στο Ισραήλ. Δυστυχία, κακομοιριά και εις βάρος των παιδιών. Τα παιδιά δεν μπορούν να, να έχουν την οσυλία που πρέπει και φύσανται κρατοριασμούς. Και το θέμα της επικοινωνίας είναι πάρα πολύ βασικό. Ούτε αυτό που μας δείχνουν τώρα μπορούμε να έχουμε καμία διαβεβαίωση ότι είναι ε, αυθεντικά. Επομένω, θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο τι πραγματικά συνέβη. Επίση, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει αυτή, να έχει αυτή την παθητική στάση, να γίνει παράγοντα διασφάλιση τη ειρήνη και θα πρέπει με ξεκάθαρα ε, αυτή τη φορά να πούμε ότι το παραέκανε το Ισραήλ και ότι θα πρέπει άμεσα να παγώσουν όλες οι συμφωνίες που έχουμε με το Ισραήλ περιμένοντας τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε διάβημα και στον ΟΟΣΑ ούτως ώστε η διαδικασία η οποία ξεκίνησε για την εισδοχή του Ισραήλ στη δημοκρατική λέσχη ε, όσων σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παγώσει επίσης, να ανασταλεί εν αναμονή της αυτής της ε, ανεξάρτητης έρευνας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Άτκινς, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Όταν πριν από 50-60 χρόνια τερματίστηκε η Βρετανική Αυτοκρατορία, βρεθήκαμε υπό πολιορκία από διάφορους ανθρώπους που θεωρούσαμε τρομοκράτες. Ο κ. Κινιάτο, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο κύριος Μπεγκίν και οπωσδήποτε τον ΑΕΡΕΗ. Τελικά αναγκαστήκαμε να τους μιλήσουμε. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ένα ηγετικό ρόλο να αναγνωρίσει τη Χαμάς, να αναγνωρίσει πως έχει σημαντικό ρόλο να παίξουν όπως είδαμε όταν πήγαμε πέρσι τον Δεκέμβριο σε μια αντιπροσωπεία εκεί πέρα. Είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι εκεί πέρα, με αυτούς πρέπει να μιλήσουμε. Επιπλέον, Μήπως είναι προφανές πλέον πως το κουαρτέτο είναι απλά μια ακριβή σπατάλη χρόνου και πως θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσουμε ότι κάτι κάνει αντί να μιλάει. Τέλος πάντων τώρα, ας μην ε, θεωρεί ότι θίγω τον κύριο Μπλερ για κομματικούς λόγους, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, μια ηγεσία και τέλος δεν αποτελεί μομφή προς το Ισραήλ το ότι μοιάζουν ανίκανοι. Έχουμε την υπερβολική αντίδραση στη Γάζα, τα προβλήματα με τα διαβατήρια, τα όσα έγιναν στην επίσκεψη Biden και τώρα αυτά εδώ πέρα, τα οποία μας δείχνουν πως χάνει την ικανότητά του, αν μη κάτι άλλο, το Ισραήλ. Και αντιλαμβάνομαι βεβαίω το πώς αισθάνεται το Ισραήλ, αλλά αν αισθάνονται υποπολιορκία θα αντιδράσουν υπερβολικά. Οπότε πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει πως θα γίνουν συνομιλίες με τη Χαμάς για να λυθούν αυτά τα δύσκολα προβλήματα και να δούμε το μέλλον των ανθρώπων της Γάζας και της Παλαιστίνης συνολικά. Ευχαριστώ Λέζινγκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω πως μου είναι δύσκολο να παραμείνω αντικειμενική μετά από αυτή την πρόκληση και το φιλμα, αυτό το φιλμάκι της προπαγάνδας. Μιλάμε για γυναίκες, ηλικιωμένους, ε, μέλη της ε, Γερμανικής Βουλής που ήταν σε αυτό το πλοίο. Τώρα το να λέει τρομοκράτες είναι για μένα προσωπική προσβολή. Ευτυχώς αυτές οι γυναίκες επέστρεψαν σήμερα και μας είπαν από πρώτο χέρι το τι γίνεται, ότι 40 άτομα ακόμα κρατούνται και δέρνονται στις φυλακές. Προσωπικά επίσης ε, διαπίστωσα πως όλες οι δηλώσεις του Κοινοβουλίου θεωρούν την περίπτωση ως λήξασα. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι φυλακισμένοι και θέλω να ακούσω πώς θα ασκηθεί πίεση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε τα άτομα αυτά να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν και να τους φροντίσουμε. Και θέλω να θέσω το ερώτημα τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους και πώς θα τους φροντίσουμε και τι, ποια θα είναι η συνέχεια. Κάτι άλλο. Λέτε συνέχεια πως στηρίζουν τρομοκράτες. Κοιτάξτε, υπήρχε αυτή η παλιά παροιμία που λέγαμε στη Γερμανία να κάνουμε τα σπαθιά άρωτρα. Αλλά αυτό το πώς θα γίνουν ε, οι αναπηρικές καρέκλες όπλα δεν νομίζω να έχει ανακαλυφθεί ακόμα αυτή η διαδικασία. Γιατί αναπηρικά καροτσάκια κουβαλούσαν οι άνθρωποι στη Γάζα. Ευχαριστώ. Μάγκλινερ eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έχω ένα σύντομο ερώτημα, αλλά θα το δούμε. Εγώ εντυπωσιάστηκα από το φιλμάκι αυτό. Βλέπεις πως πάλευαν για τη ζωή τους οι στρατιώτες. Και ε, ναι. τώρα οι ειρηνιστές, τι ειρηνιστές, οι ειρηνιστές δεν υποδέχονται τους στρατιώτες με ρόπαλα. Το, το, το είδατε τι έγινε. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι Ε, έπεσαν όντως ε, νεκροί κατά τη διάρκεια αυτής της, ε, της αυτοάμυνα, γιατί είναι σαφές πως ε, ήταν σε αυτοάμυνα. Ευχαριστώ. Ο πρέσβης ο κύριος Κούριελ για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Οπωσδήποτε θα μεταφέρω στην κυβέρνησή μου την εντύπωση που αποκόμισα από αυτή τη συνεδρίαση και αυτά τα οποία είπε ο κάθε ένας εδώ μέσα. Να ξεκινήσω ίσως από την πλευρά Ισραήλ-Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απαντήσω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βίγκελ για την επίσκεψη. Ο τίτλο. δεν ξέρω. Ίσως να είναι τεχνικό πρόβλημα. Ο τίτλο ήταν παραπλανητικό γιατί έλεγε «Επίσκεψη στο Ισραήλ και στι Παλαιστινιακέ περιοχές» και ε, ήταν επίσκεψη στι Παλαιστινιακέ περιοχές. Μόνο. Και ε, ασχολήθηκαν με το Ισραήλ μόνο υπό το πρίσμα των Παλαιστινίων. Δηλαδή, πήγατε στους Παλαιστίνιους και μετά ήρθατε να συναντήσετε με το, το Ισραήλ για να μιλήσετε μόνο για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Θέλετε να δείτε το Ισραήλ, ελάτε. Δείτε την οικονομία του Ισραήλ, την κοινωνία των πολιτών, την νεολαία. Δεν μπορείτε να μεταμορφώσετε την ε, σύγκρουση αυτή στο μόνο ζήτημα που θα απασχολεί το Κοινοβούλιο σας. Γνωρίζω πως είναι σημαντικό, αλλά αν θέλετε ε, να σας παίρνουμε σοβαρά στο Ισραήλ, πρέπει να έρθετε σε επαφή με το Ισραήλ αντί να μας κάνετε μόνο μάθημα και καταδίκη. Το παρατήρηση. Δεύτερη. Δεύτερον, το Ισραήλ πράγματι θα κάνει τις σωστές έρευνες. Το κάνουμε κάθε φορά. Ήταν αναπάντεχο αυτό το αποτέλεσμα. Δεν περιμέναμε να έχουμε θύματα σε αυτή την επιχείρηση και δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα ερευνήσουμε και για, για, για μας. Όχι για το χατήρι κανενός εκτός του Ισραήλ. Προς την κυρία Ζολή αναφέρατε την ιατρική κατάσταση στη Γάζα. Δεν. Μου φτάνει τώρα ο χρόνος να αναφερθώ στις συνολικές σχέσεις Γάζας και Ισραήλ, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται ιατρικός διάδρομος. Μόνο το 2009, 10.000 άνθρωποι από τη Γάζα έτυχαν ιατρική περίθαλψης στο Ισραήλ. Υπάρχει λοιπόν ένας διάδρομος για να φεύγουν οι ασθενείς από τη Γάζα και 200, 200 ε, άτομα ιατρικό προσωπικό μπαίνουν βγαίνουν κάθε μέρα. Επίσης, 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο ξοδεύονται για την περίθαλψη Παλαιστινίων στο Ισραήλ. Δεν είμαστε αδιάφοροι στον πόνο που υφίσταται στην Γάζα. Αλλά υπάρχουν και άλλα διλήμματα. Όσον αφορά τη Χαμάς. Δεν μπορείτε να πείσετε τη Χαμάς να αποδεχτεί τα βασικά κεκτομένα, κεκτημένα της ειρηνευτικής διαδικασίας. Τι ζητάμε, αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ να υπάρχει. Δηλαδή μιλάμε για λύση δύο κρατών. Αλλιώς δεν υπάρχει ποτέ άλλο να συζητήσουμε. Εάν η θέση της Χαμάς παραμένει πως το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει και μιλάμε για ένα κράτος Παλαιστινιακό, δεν έχει τίποτα να ζητήσουμε. Δεύτερον, να αποκηρύξει βία τι πιο βασικό από αυτό. Και τρίτον, να αποδεχτεί τις προηγούμενες συμφωνίες για να μην ξεκινάμε από το μηδέν. Εάν πείσετε τη Χαμάς για αυτά τα τρία στοιχεία, θα διαπραγματευτούμε μαζί τους. Ε, δεν ελπίζουμε εσείς να διαπραγματευτείτε μαζί τους, εμείς θα τους μιλήσουμε. Το ερώτημα δεν είναι να μιλήσουμε ή να μην μιλήσουμε με τη Χαμάς, αλλά το τι θα συζητήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να τηρήσετε τις αρχές του κουαρτέτου, κάτι το οποίο δεν κάνετε αν δείτε τα τελευταία συμπεράσματα και δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, πριν από δύο χρόνια δεν υπάρχουν. Η Χαμάς θεωρεί πως κερδίζει δηλαδή. Μπορεί να συνεχίσει η τρομοκρατία και ο ένας αποκλεισμό ή ο άλλος θα σπάσει τελικά και θα κερδίσουμε. Αυτά είναι βασικά τα σχόλιά μου. Από την άλλη είμαι διατεθειμένο να, να παραμείνω σε επαφή μαζί σα και με το Κοινοβούλιο. Το, το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να παραμείνει σε επαφή μαζί σα. Με κατηγόρησαν πω δεν ήρθα στη συνεδρίασή σας την τελευταία φορά πριν πάτε στο Ισραήλ. Δεν με προσκάλεσαν ποτέ. Εάν με είχαν προσκαλέσει, ευχαριστώ, θα είχα έρθει και θα σα εξηγούσα πώ θα γίνονταν πιο ισορροπημένο αυτό το πρόγραμμα από ό,τι ήταν ε, στα χαρτιά. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να με προσκαλέσουν, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Στο σημείο αυτό νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε την συζήτηση. Αλλά έχουμε εδώ πέρα 18 συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν. Και έχει τελειώσει ο χρόνος με διερμηνία, οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω τα σχόλιά σας να περιοριστούν σε ένα λεπτό και αν θέλετε να μας πείτε σε ποιον απευθύνονται τα σχόλιά σας. Και τώρα θα δώσουμε λόγο στον ε, ένα ή στον άλλο ε, πρέσβη, ανάλογα με ποιον ρωτήσετε, και τώρα κύριο Φιδεκτήση το λόγο για ένα λεπτό. Κασουλίδη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε για αυτό το λεπτάκι που το οποίο μου έχετε δώσει, θέλω πρώτα-πρώτα να ρωτήσω τον πρέσβη, τον κύριο Φερνάντε. Όταν μιλούμε για μια πλήρη και ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα υπό ποιο θα γίνει αυτή το γεγονό ότι έγινε σε διεθνή ύδατα το επεισόδιο. Αυτό δικαιολογεί το Ισραήλ να διεξαγάγει αυτήν την έρευνα ή θα είναι διεθνής αυτή η έρευνα και θα είναι δυνατόν να κλητευθεί οποιοδήποτε από του εμπλεκομένου ούτω ώστε να προσέλθει να καταθέσει. Τώρα μια δεύτερη ερώτηση η οποία αφορά τον Ισραηλινό πρέσβη, τον οποίο ευχαριστούμε που άμεσα κινητοποιήθηκε για να έρθει εδώ. Θα ήθελα να μου πει για το κατά πόσο είναι δυνατόν έχουμε μια πολιτική λύση στο πρόβλημα του αποκλεισμού. ταυτοχρόνω δε πώς θα γίνει να σταματήσει το λαθρεμπόριο των όπλων. Ανεξαρτήτως και πέραν του τι κάνει, τι δεν κάνει η Χαμάς. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Κασουλίδη και τώρα η κυρία Κοπάχη το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε. Η χθεσινή αιματηρή επίθεση Ισραηλινών κομμάτων εναντίον της Ειρηνική νιοπομπής που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό στη Γάζα σε διεθνή ύδατα αποτελεί ένα πρωτοφανές γεγονός, μια πράξη πειρατείας. Ο θάνατος και ο τραυματισμός ειρηνικών ακτιβιστών που με αυταπάρνηση προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους κατοίκους της Γάζας είναι γεγονότα παράδεκτα που προσβάλλουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου ή διεθνού τάξης. Περιμένουμε απαντήσει, και αυτέ τι απαντήσει δεν θα μα τι δώσει έρευνα από πλευρά του Ισραήλ όπω πρότεινε χθε η Βαρόνι Άστο στο πρώτο ανακοινοθέν τη, το οποίο ευτυχώ ε, διόρθωσε. Απαιτείται ισχυρή καταδίκη των ενεργειών αυτών του Ισραήλ, άμεση λύση του αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων και πάγωμα της Συμφωνίας Σύνδεσης έως την πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση της υπόθεσης σε κάθε περίπτωση να δούμε με αρμόζουσα σοβαρότητα το δράμα του πληθυσμού της γάζας και συνάδελφοι δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. κανείς δεν είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου. ευχαριστώ. Ε, για ένα λεπτό. My apologies. Συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, νόμιζα πως είχε τελειώσει ο κατάλογος των ομιλητών, οπότε είχα άλλη δουλειά. Αναρωτιόμουν εάν ο κύριος πρέσβης μπορεί να μας εξηγήσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν όταν προσπάθησαν να αλλάξουν ε, πορεία στο στόλο, στο στολίσκο, και ποιος έλαβε την απόφαση επιβίβασης στα, στα πλοία, γιατί φαίνεται πως ε, υπήρξε μια πρώτη βίαιη επαφή και αναρωτιόμουν ποια άλλα μέτρα ελήφθησαν πριν από αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ. Ο κ. Στοημόπουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι υποστηρίζω τη συνύπαρξη και τις μη βίαιες λύσεις. Όμως αυτό που ακούσαμε για βίαιο και προκλητικό στο Λίσκο στην πράξη μετέφερε τρόφιμα, φαρμακευτικό και οικοδομικό υλικό. Υπάρχουν αποδείξεις από την έρευνα ότι μετέφερε κάτι άλλο. Επειδή κρατούνται παράνομα οι ειρηνιστές και οι υπόλοιποι γίνονται αντικείμενο κακομεταχείρισης, ακούσαμε τον ένα καπετάνιο να καταγγέλει ξυλοδαρμό του συντονιστή της αποστολής που έχει το όνομα Βαγγέλης Πισίες. Ένα άλλο μέλος του πληρώματος κατήγγειλε ότι γίνεται ηλεκτροσόκ. Θα ήθελα να σχολιαστεί από την Επιτροπή η εξή πρόταση, οι προτάσεις. Να καταστήσει υπεύθυνο το Ισραήλ για την υγεία των απαχθέντων, να ζητήσει την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωσή τους και αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάει άμεσα με αεροπλάνο και ιατρική υποστήριξη για να παραλάβει τους απαχθέντες που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί με άγνωστες συνθήκες και χωρίς επικοινωνία. Κύριε Πρόεδρε, είναι βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε την αξιοπιστία του μηχανισμού που μόλις μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε φτιάξει για να ασκήσουμε μια σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πρέπει να κινηθούμε σε τέσσερις κατευθύνσεις. Ανεξάρτητη διερεύνηση του συμβάντος. Μια ισχυρή πρωτοβουλία για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας μια επανεκκίνηση της, δια... της ειρηνευτικής διαδικασίας, συνομιλώντας με όλους όσους μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Και βεβαίως να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση για το πώς θα προχωρήσουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ. Έχω τρεις ερωτήσεις για τον, πρέσβη, για τον αξιότιμο κύριο Πρέσβη. Για το φιλμάκι που είδαμε. Είπατε ότι είχατε πληροφορήσει ότι υπήρχαν όπλα. Για αυτά τα όπλα μας μιλάγατε. Αυτά τα όπλα έχει ανάγκη η Χαμάς αυτή τη στιγμή. Αυτά τα όπλα θα έδιναν στους τρομοκράτες. Τι περιμένανε να τους υποδεχθούν οι στρατιώτες που κατέβαιναν με λουλούδια. Προφανώς όχι. Το πρόβλημα κύριε Πρέσβη είναι ότι τα ρόπαλα φαίνονται, οι σφαίρες όχι. Bene, onorevole Tannock, ecco, toccherebbe a lei <laughs> se si porta Ε, μια, περισσο... μια διευκρίνηση. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο, δεν θα πρέπει να κατηγορούμε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κατασκευάζει αποδείξεις, αυτό είναι ανοησία. Η ερώτησή μου νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι πληροφορίες χθε έλεγαν ότι βρέθηκαν δύο περίστροφα σε ένα πλοίο και ότι ένα όπλο αφαιρέθηκε από ένα Ισραηλινό στρατιώτη και μετά χρησιμοποιήθηκε εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ. Μπορεί να το επιβεβαιώσει ο πρέσβης αυτό. Χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου είδους πειρά ε, εις βάρος των Ισραηλινών στρατιωτών. Ευχαριστώ. Κέλα με ένα λεπτό. οπότε ο κύριος Στρίφλερ, για ένα λεπτό. Ναι κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να πω ότι αυτά τα οποία λέγατε προηγουμένως με εντυπωσίασαν. Μιλήσατε στους ευρωβουλευτές και είπατε ότι αν θέλετε το Ισραήλ να πάρει σοβαρά αυτά που λέμε. Αν θέλετε εμείς να πάρουμε σοβαρά αυτά τα οποία εσείς λέτε θα πρέπει να πάψετε να απαγορεύετε την είσοδο των και ευρωβουλευτών στη Γάζα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εγώ πήγα στη Γάζα, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι που ήταν μαζί μου, συναντήσαμε την απόλυτη φτώχεια. Θα ήθελα να πω επίσης κύριε Πρέσβη ότι το Χαμάς τροφοδοτείται από το Ισραήλ γιατί μέσω αυτού του, ε, αυτού του αποκλεισμού ωφελείται πολιτικά το Χαμάς. Καιρός είναι λοιπόν να σπάσετε αυτόν τον αποκλεισμό. Τελειώνοντας, να υπογραμμίσω ότι συνάντησα την Ιερουσαλήμ μια Ισραηλινή η οποία μου είπε ότι ντρέπεται για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση γιατί η πολιτική αυτή δεν υποστηρίζεται από όλο το λαό του Ισραήλ. Σίβια και ένα λεπτό. Ε, ε, Είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάει κανείς ε, έμφορτο συναισθηματικά. Το θέμα είναι ότι είδαμε αίμα ε, στις εικόνες της τηλεόρασης και αυτό είναι τρομερό και θα πρέπει με ψυχραιμία σαν πολιτική υπεύθυνη να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Οι θέσεις του Συμβουλίου με βρίσκουν σύμφωνο. Και εκφράζω την ικανοποίησή μου για την αντίδραση της υπηρεσίας της κυρίας της οποίας προείσταται η κυρία Άστον. Εμείς προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με ειρηνικό τρόπο. Το θέμα είναι βέβαιο ότι κάποιος έχει πολεμικές διαθέσεις θα έλεγα. Κάποιος έβαλε όλους αυτούς τους ανθρώπους στα πλοία και τους οδήγησε σε αυτήν την περιοχή που βρίσκεται σε πολεμική κατάσταση και έτσι προκλήθηκε αυτή η τραγωδία. Και κάποιος έδωσε επίσης μια ανόητη διαταγή στους Ισραηλινούς στρατιώτες να πυροβολήσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν, ε, είναι ικανο... δεν ε, ήταν ένοπλοι. Εν πάση περιπτώσει. Έχουν ε, προκληθεί πάρα πολλά προβλήματα, όλοι είναι δυστυχείς από αυτό το οποίο συνέβη και ο μόνος ευτυχής σε αυτή την περίπτωση ήταν ο υπουργό του Ιράν, ο οποίος εποφελήθηκε το συμβάν το τραγικό και εξέφασε αυτές τις απόψεις που ακούσαμε. Η κυρία Θεοχάρου dalle 6.45 Από 6 και 45 μέχρι τις 7 βεβαίως δεν θα έχουμε όλες τις γλώσσες. Θα μπορείτε να μιλήσετε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Πέρυσι στις 29 Δεκεμβρίου του 2008, με συγχωρείτε, ήμουνα επάνω στο μικρό πλοίο Dignity, 10 φορές πιο μικρό από το Μαβί Μαρμαρά, και κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Γάζας, ξεκινήσαμε να μεταφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ε, για να, πιο πολύ για να στείλουμε και διάφορα μηνύματα και προς τον λαό της Γάζας και προς το Ισραήλ και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας βυθίσατε 70 ναυτικά μίλια δυτικά της Χάιφας, το πολεμικό σας ναυτικό, και μας έσωσε το γαλλικό ναυτικό. Ελπίζω ότι θυμάστε αυτή την ιστορία. Μα είπατε πριν από λίγο ότι μπαίνουν συνέχεια όπλα στη Γάζα από, πολεμικά, από, από, από τη θάλασσα. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξή. Γιατί πάντα επιτίθεστε εναντίον πλιαρίων εθελοντών και ποτέ δεν σας ακούσαμε να επιτίθεστε εναντίον πλιαρίων που μεταφέρουν όπλα. Ένα ερώτημα. Δεύτερο, πώς είναι δυνατόν τα πιο καλά σας κομάντο να αφοπλιστούν από ανθρώπους που ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα. Και τρίτο, μια ερώτηση για την Κομισιόν. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, την επαύριο που βυθίστηκε τον Τίγνητη, την επαύριο που βυθίστηκε τον η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εισηγήθηκε, η Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα, εισηγήθηκε να ανοίξει ένα θαλάσσιο διάβλο προ τη Γάζα και αποφασίστηκε αυτή η υπόθεση. Φαντάζομαι ήταν μια ανάλογη ιστορία με τώρα. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Σα ευχαριστώ. Ονορεύολε Τάλερ, per Τάλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχολείο μου αφορά τον κύριο Πρέσβη. Είπε πως θα τα μεταδώσει όλα προς την κυβέρνησή του. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο εμείς οι φίλοι του Ισραήλ πρέπει να προστατεύσουμε το Ισραήλ από τον εαυτό του. Η Γάζα έχει καταντήσει συνώνυμο του γκέτο μέσω της Ισραηλινής πολιτικής σαν το γκέτο της Βαρσοβίας, του Σαράγεβο και τα λοιπά. Τα γνωρίζαμε όλα αυτά. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι, οδηγεί σε εντάσεις η εμπλοκή μας δηλαδή. Αυτό εδώ πέρα η πράξη θα δημιουργήσει περισσότερους τρομοκράτες από όσους μπορεί να παρεμποδίσει το Ισραήλ και εμείς κοιτάμε πρέπει να κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο παρατηρητές. Πρέπει να βοηθήσουμε το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους να ιδρύσουν ένα κράτος της Παλαιστίνης που θα υπάρχει δίπλα στο Ισραήλ και να το προστατεύσουμε για να ζήσουν ειρηνικά οι επόμενες γενιές. Αυτή είναι η αποστολή μας. Σας ευχαριστώ. Φλότρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τέλος πάντων δεν θέλω τώρα να ξεκινήσει μία νέα συζήτηση προπαγανδιστική η οποία θα είναι ανάξια μας. Θα ήθελα απλά να θέσω ένα απλό ερώτημα κύριε Πρέσβη. Γνωρίζετε τον αριθμό των ατόμων που σκοτώθηκαν και τον αριθμό των ατόμων που τραυματίστηκαν σε αυτό το περιστατικό. Σκοπεύετε να εκφράσετε συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και θα μπορούσε ίσως να προταθεί ε, να τηρήσει ενός λεπτού σιγή η Κνεσέτ για αυτά τα θύματα, για τα δε άτομα που κρατούνται στο Ισραήλ. Πώς θα μπορέσουν να σκίσουν τα δικαιώματά τους, να απολαύσουν τις ελευθερίες τους, θα μπορέσουν να πάνε στην Γάζα. Θα επιτρέψετε μία μερόληπτη διεθνή έρευνα και σκοπεύετε να ζητήσετε από την κυβέρνησή σας μετά από αυτή την συζήτηση να σεβαστεί το Ισραήλ τις συμφωνίες που έχει υπογράψει ειδικά όσον αφορά την διακοπή του προγράμματος ε, των ε, επικισμών. Ε, είστε πολύ αυστηρός κύριε Πρόεδρε, τώρα για 10 δευτερόλεπτα είμαι με όλους λέει ο κύριος Πρόεδρος. και για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν λέμε για άμαχους και για πολίτες, είναι εκείνοι που έπεσαν θύματα της επίθεσης των στρατηγών και ε, λέμε και για ε, αυτούς που υποφέρουν στη Γάζα το και τότε χτυπάει η καρδιά μας πιο δυνατά και επομένως γι' αυτό και εμείς θέτουμε αυτά τα ερωτήματα όσον αφορά τους λόγους, τις αιτίες ε, δεν πρέπει να είμαστε μονοπλευροί, αλλά καμιά φορά είμαστε μονοπλευροί. Γινόμαστε μονοπλευροί γιατί καθόμαστε και, και, και σκεφτόμαστε αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί τόσες, τόσες επιθέσεις. Και, αλλά από την άλλη μεριά φυσικά και η Χαμάς έχει κάνει επιθέσεις. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, να μπούμε στην ουσία του θέματος. Γιατί ούτε η Χαμάς ε, σέβεται το δικαίωμα του Ισραήλ το να υπάρχει και το Ισραήλ δεν σέβεται τα δικαιώματα των κατοίκων της Γάζας. Έχουμε την Τουρκία που είναι ο εταίρος μας, ο συνομιλητής μας στην περιοχή και μπορεί η Τουρκία να βοηθήσει, μπορεί να ασκήσει πίεση στη Χαμάς αλλά και στο, και, Ιράν που βρίσκεται πίσω από, από τη Χαμάς. Κύριε Πρέσβη, φαντάζεστε πώς μπορεί να ασκείτε κριτική στις πράξεις κυβέρνησής σας και ταυτόχρονα να υπερασπίζεστε το δικαίωμα υπέρ του Ισραήλ. Δεύτερον, είστε σε κατάσταση ένοπλη σύγκρουση με τη Χαμά, γιατί αυτό έχει συνέπειε όσον αφορά τον ε, ναυτικό αποκλεισμό. Επίση, όσον αφορά την παρέμβαση. Υπάρχουν διάφορα τμήματα στην κλιμάκωση. Μπορείτε να προσπαθήσετε να χτυπήσετε την πλώρη του πλοίου τα κτλ. Ισχύει επίσης πως πυροβόλησαν από τα ελικόπτερα από αέρος η Ισραηλινοί στρατιώτες. Επίσης, συμφωνείτε, θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνής ανεξάρτητη επιτροπή έρευνα και όχι μια Ισραηλινή. Πρέντα για ένα λεπτό. Δεν είναι εδώ, ντερόσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, έχω ένα ερώτημα για τον κύριο πρέσβη του Ισραήλ. Θα συνεργαστεί το Ισραήλ με μια διεθνή έρευνα εάν υπάρξει τέτοια. Ε, καθώς δεν είχε συνεργαστεί με την έρευνα Goldstone. Θα αναγνωρίσει επίσης πως είμαστε επιφυλακτικοί για το βίντεο που μας έδειξε. Όχι γιατί ξέρουμε τι είναι το σωστό ή το λάθος, αλλά γιατί ο κύριος Ντανιέλ Τάουμπο επικεφαλής, ένας από τους επικεφαλής. Ε, συνομικού συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών μας έδειξε κάποιες εικόνες πριν την έκθεση Γκολτσόν που αποδείχθηκε πως δεν είχαν σχέση με τη συγκρούστη Γάζα αλλά ήταν από το 2004, 5 και 6. Οπότε είμαστε επιφυλακτικοί για εικόνες που μας δείχνετε εκτός εάν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του. Και τέλος να σας πω πώ. το βασικό θέμα εδώ πέρα σχέση με τη Χαμά είναι πως θα πρέπει να δεσμευτούν πως δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ βία για να επιτύχουν τους σκοπούς τους ανεξαρτήτως αγνώριση του Ισραήλ. Αυτό έκανε και ο IRA και μέχρι τώρα ποτέ δεν έχει αποδεχτεί την νομιμότητα της αγγλικής κυριαρχίας στη Βόρεια Ιρλανδία αλλά δεσμεύσει και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία.